Ο πρόεδρος Μάρτιν Σούλτ. κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, σα παρακαλώ καθίστε, αρχίζει η συνεδρίαση. κυρίε και κύριοι, αξιότιμες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για μια ιστορική πρόκληση. Αυτή είναι που αντιμετωπίζουμε με το κύμα των προσφύγων. Χρειάζεται αλληλεγγύη και προς τα μέσα και προς τα έξω. Γι' αυτό και θα ψηφίσετε αμέσως τώρα για ένα κατεπήγον μέτρο για την